Ah, j'adore ce marteau. Hein. <laughs> si vous voulez prendre place, s'il vous plaît. Καθίστε παρακαλώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους σας. Ε, ε, A Και ελπίζω η χρονιά αυτή να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Κατόπιν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Προέδρου μας, του κ. Βόμποντα, που δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα. Και Αναλαμβάνω λοιπόν καθήκοντα εγώ. Έχουμε αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 25 θα γίνει αμέσως μετά το σημείο 9. Το 24 θα γίνει μετά από το σημείο 16. Και τα σημεία 5, 12, 13, 14, 17, 18 και 20 αναβάλλονται. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση λοιπόν εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να έχετε μαζί σας τις κάρτες σας για την ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν ε, δεν υπάρχει αντίρρηση, μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά Τη συνεδρίαση τη 28 η και 29 η ε, Νοεμβρίου και της 17 η Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Πνευματικά δικαιώματα στην ε, ψηφιακή ενία αγορά και να δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Κομοντίνη, η οποία είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Μπελβό. Καλημέρα σε όλους και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά. Η συζήτηση για αυτή την οδηγία ξεκίνησε πολύ γρήγορα. Έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις με τους ε, ενδιαφορομένους. Εδώ στην Επιτροπή ε, κάναμε και δημόσια κρόαση και είχαμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποιες από τις πτυχές ε, των προτάσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την ακρόαση. Δεν ε, θα ήθελα να σας καθυστερήσω πολύ. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να ακούσω τις ε, θέσεις ε, των σχεδόν εισηγητών και τυχόν θέματα που τους απασχολούν. Η γραμματεία ε, με βοήθησε να καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα και έχει δημοσιευθεί και όλας. Συνεργαζόμαστε βεβαίως και με την Επιτροπή ΙΜΚΟ επ' αυτού. Θα μας δώσουν και αυτή τη θέση τους. Η Επιτροπή Πολιτισμού ζήτησε επίσης ε, να ε, γνωμοδοτήσει επ' αυτού και έχουμε σχεδόν καταλήξει σε συμφωνία για ε, την ε, γνωμοδότησή τους. Ε, νομίζω ότι και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έστειλε έτοιμα στη Γραμματεία για να υποβάλουν και αυτή την άποψή τους. Ε, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πρόβλημα να λάβουμε γνωμοδοτήσεις από οποιαδήποτε Επιτροπή, αλλά έχω αρχίσει και ανησυχώ επειδή ακριβώς πρόκειται για θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι ένα θέμα που αφορά κυρίως ε, πνευματικά δικαιώματα και ο κανονισμός προβλέπει ότι τα πνευματικά δικαιώματα εμπέπτουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Αρκετέ αρκετές άλλες όμως επιτροπές ζήτησαν άρθρο 54. Και εδώ ανησυχώ λίγο, διότι δεν θα ήθελα η Επιτροπή να βρεθεί ε, και ενώπιον ε, αμφιλεγόμενων και διστάμενων θέσεων. Όπως σας είπα, έχω ακολουθήσει μια πάρα πολύ διάφανη διαδικασία. Όλες οι πληροφορίες των συνεδριάσεων που κάνουμε τους ενδιαφερομένους ε, διατίθενται δημοσίως ε, στο διαδίκτυο. Ακόμα και οι ακροάσεις της δικής μου πολιτικής ομάδας ήταν ανοιχτές προς το κοινό. Και όταν συναντώ συναδέλφους ε, με αρκετές ε, πολιτικές ομάδες, αλλά ε, το να υπάρχει δυνατότητα άρθρου 54 σε άλλες επιτροπές με ανησυχεί. Όχι μόνο γιατί τα πνευματικά δικαιώματα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, αλλά γιατί μπορεί να καταλήξουμε σε ιδιαίτερα διστάμενες θέσεις σε ένα ε, θέμα το οποίο ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλές διαφορετικέ απόψεις ε, μεταξύ των ενδιαφερομένων. Αυτά λοιπόν τα περί επιμελητίας του ζητήματος. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν κάποιες πτυχές οι οποίες θα έλεγα ότι σίγουρα αποτελούν αντικείμενο περισσότερες συζήτηση και μεταξύ των συναδέλφων και μεταξύ των ενδιαφερομένων. Και αυτά είναι κυρίως το άρθρο 11 και το άρθρο 13 τα δικαιώματα των ε, ε, εκδοτών και η σχέση που υπάρχει μεταξύ της κάθε πλατφόρμας και αν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε ευθύνε ε, για περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες που μπορεί να δημιουργήσει θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου εν είδη γενική εισαγωγή και φυσικά προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και ε, είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω όλες τις απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάσα και πρέπει να πω ότι αντιλαμβάνουμε και την ανησυχία σου για τη συνεργασία με τις άλλες επιτροπές. Δεν είναι πάντα πολύ εύκολη συνεργασία. Να δώσω πρώτα το λόγο στη Λίντια και κατόπιν η Τζούλια και η Μέρη. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και για τη χθεσινή συνεδρίαση, η οποία ήταν άκρος ενδιαφέρουσα. Ιδίως διότι ακούσαμε εντελώς διαφορετικές απόψεις για ένα αρκετά επίμαχο θα έλεγα ζήτημα στο πλαίσιο της Επιτροπής μας διότι πρόκειται για τα δικαιώματα δημιουργού, τα πνευματικά δικαιώματα. και το λεγόμενο value gap, ένα αξιακό χάσμα. Υπάρχει λοιπόν ε, πολλή συζήτηση γύρω από όλο αυτό το θέμα που είναι αρκετά αμφιλεγόμενο και κατά την άποψή μου δεν είναι κάτι αναγκαίο δυνάμει του νέου κανονισμού. Ζούμε σε έναν κόσμο που οι συμπολίτε μας χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις πολιτιστικέ υπηρεσίε διαβάζουν περισσότερα βιβλία, εφημερίδε. Αυτό διότι έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε τέτοιο υλικό. Υπάρχουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες, το Google για παράδειγμα. Χθες ε, μάλιστα λάβαμε απευθείας ενημέρωση από το διευθυντή της Google. Εν λόγω πλατφόρμες με πολύ διαφανή τρόπο παρουσιάζουν τα κέρδη που αποκομίζουν από τη διάθεση αυτού του επιγραμμικού περιεχομένου ή το ότι μπορούν να παραπέμπουν τους ενδιαφερομένους στο περιεχόμενο αυτό. Το ίδιο και για τους εκδότες. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που δημιουργούν πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Οι εκδότες, σε περισσότερες περιπτώσεις, έχουν δικαιώματα δημιουργού. Αυτό είναι άλλωστε προϋπόθεση συνεργασίας για την έκδοση ή για την πρόθεση ενός έργου. Στο άρθρο 11 συγκεκριμένα έχουμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Κατά την υπόψη μου, δεν χρειάζεται να περιπλέξουν περαιτέρω τα πράγματα στο σημείο αυτό. Υπάρχει επίσης πολλή συζήτηση γύρω από το γεγονός ότι πρόκειται για δικαίωμα με αναδρομική ισχύ, δηλαδή μπορούμε να γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω. Ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε καν μορφή του που έχει σήμερα αυτό το έργο. Και σίγουρα δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, δεν έχουν διασαφιστεί επαρκώς. Έχουν και το άρθρο 15 Μπορούμε μεν να συμφωνήσουμε ως προς το ότι η οδηγία κατά κάποιο τρόπο ενισχύει τη θέση των δικαιούχων, των κατόχων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τους ως πληρωμής, αμοιβή. Οι προτάσεις είναι πολύ σαφέστερες ε, και εξασφαλίζεται πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί. Όμως, εγώ στην πράξη πώς θα λειτουργήσει δεν το κατανοώ, όσο και αν είναι ξεκάθαρο το σύστημα. Άρα, ναι, μεν καλές προθέσεις υπάρχουν, η πραγματικότητα όμως θα είναι πολύ δύσκολη για να τα αποκρισταλώσουμε όλα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό. Άρα η πρόταση δεν είναι καλή κατά την άποψή μου, διότι για μια ακόμη φορά δεν είναι ξεκάθαρο πράγματα, άρα δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Έρχομαι στο άρθρο 5. Εξαιρέσεις. Στο μέτρο του δυνατού. Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να υπάρχει εναρμόνιση των εξαιρέσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι καλύτερο σημαντικό είναι να εφαρμοστεί τάχιστα η συνδίκη του Μαρακές. Προβλέπεται επίσης ελευθερία του πανοράματος. Δεν χρειάζονται λοιπόν επιπλέον φραγμοί για επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές κτλ. γενικά για το επιστημονικό έργο. Στην πρόταση αυτή δυστυχώς φοβούμε ότι οι περιορισμοί που προβλέπονται, που είναι περαιτέρω περιορισμοί από που ήδη ισχύουν, θα δημιουργήσουν προσκόμματα και είναι κάτι απευκταίο. Δεν θέλουμε να περιπλέξουμε αντί να απλουστεύσουμε την κατάσταση. Εξάλλου σε κάθε χώρα ισχύουν διαφορετικές πραγματικότητες. Αν οι εξαιρέσεις αντιμετωπίζονται διαφορετικά, η ενιαία ψηφιακή αγορά θα είναι κάτι άκρος πολύπλοκο να επιτευχθεί παρότι είναι και η βάση της πρότασης της Κομισιόν, ακριβώς αυτή είναι η ψηφιακή αγορά. Αυτό έχω να πω στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και για τη χθεσινή συνεδρία στην άκρο ενδιαφέρουσα, όπως προείπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τον διαφανή τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί το θέμα, τις διαβουλεύσεις, τις συζητήσεις, τις ανταλλαγές απόψεων που έχουν ήδη γίνει. Βοηθά αυτό στο έργο μας επί αυτού του πολύ περίπλοκου φακέλου. Δεσμεύομαι και εγώ να συμβάλλω επικοδομητικά για να ολοκληρώσουμε αυτό το φάκελο εντό τη θητεία μα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω και εγώ ότι χρειάζεται να γίνει λεπτομερή συζήτηση για όλα τα άρθρα τη πρόταση. Η πρόταση αυτή έχει ήδη δημιουργήσει ε, διάφορες ε, και η συγγήτρια επισήμανε και τα δύο ε, πλέον αμφιλεγόμενα και επίμαχα άρθρα, τα 11 και 13, ε, πρέπει να γίνει συζήτηση όμως και επί των υπόλοιπων άρθρων ε, σε βάθος, όχι μόνο σε αυτά. Η αρχική πρόταση της μεταρρύθμισης των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως είχε ανακοινώσει τουλάχιστον ε, η, Κομισιόν, ε, απλοποίηση και η εναρμόνιση των κανόνων δεν έχουν ε, επιτευχθεί ακόμη και πιστεύουμε εμείς ως σοσιαλιστές ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να ε, εξασφαλίσουμε ότι τα μη ε, επίμαχα αιτήματα και όχι ιδιαίτερα περίπλοκα αιτήματα του κοινού, όπως είναι αυτή η ελευθερία παρονάμανση, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο. Όσον αφορά τα περισσότερο επίμαχα σημεία, άρθρα 11 και 13, πιστεύω ότι το 13 και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις δημιουργούν σύγκρουση με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία ακριβώς γιατί δημιουργούν μια άμεση ευθύνα Δηλαδή, θα ε, ευθύνονται οι ε, host providers, οι πλατφόρμες για το περιεχόμενο το οποίο ε, ανεβαίνει στις πλατφόρμες αυτές. Αυτό νομίζω ότι αντικείται στη βασικότερη αρχή που διέπει ε, τη λειτουργία του ίντερνετ από την αρχή ε, και την αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα που ε, αναπτύσσεται στο διαδίκτυο. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από ασυνέπειες, το, το ανέφερε και το EPRS, ε, ανάμεσα στην ε, εν λόγω πρόταση της Κομισιόν αλλά και την υφιστάμενη ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θέλω να σημειώσω ότι, ότι η τεχνολογία ταυτοποίησης οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικού δικαιώματος δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες, κάποια ηχητικά αρχεία τα οποία θα μπορούσαν για παράδειγμα πράγματι να εντοπίζονται από software αλλά δεν μπορεί κάτι τέτοιο να διευρυνθεί και να επεκταθεί σε όλα τα είδη περιεχομένου. Ε, συμφωνώ επίσης ε, με τα ζητήματα που έχουν θέσει άλλοι συνάδελφοι από την ε, ε, από την πολιτική ομάδα των σοσιαλιστών. Πρέπει επίσης όσον αφορά τουλάχιστον την, τα ιδιοσιογραφικές, τις πλατφόρμες. Όσον αφορά την ε, ελευθερία κυκλοφορίας και τον πλουραλισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, πιστεύω ότι το δικαίωμα να δημιουργεί κανείς συνδέσμους σε ειδήσει είναι σημαντικό να διατηρηθεί. Υπάρχει διαφορά μεταξύ, ε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα, στα πνευματικά δικαιώματα και στο, στα συγγενικά δικαιώματα. Ε, η Κομισιόν έχει ήδη αναγνωρίσει ότι αντιγραφή μιας ε, επικεφαλίδας, ε, μιας είδηση, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελεί στο μέλλον παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτό φυσικά αποτελεί πρόβλημα για την ελεύθερη κυκλοφορία ειδήσεων στο ίντερνετ. Επίσης, πολλές φορές το περιεχόμενο ε, δεν είναι σαφές από έναν τίτλο είδηση που μπορεί να δει ένας ε, χρήστης. Ε, γι' αυτό είναι παράλογο να ζητείτε από μια πλατφόρμα να καταβάλει δικαιώματα ή αμοιβέ απλά και μόνο διότι χρησιμοποιεί ορισμένους όρους ή συγκεκριμένες λέξεις. Αυτά ως προς τα συγγενικά δικαιώματα. Για παράδειγμα υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ένα τραγούδι και ένα ηχητικό αρχείο ε, ενώ τα κείμενα ε, είναι ε, πραγματικά εντοπίσιμα αν έχουν πράγματι αντιγραφή. Κατά τη γνώμη των σοσιαλιστών λοιπόν θεωρούμε ότι τα άρθρα 11 και 13 πρέπει να διαγραφούν και αντιθέτως θα πρέπει να αντικατασταθούν από προτάσεις που θα απλουστεύουν και θα εναρμονίζουν τους κανόνες. Άλλες, ε, άλλα στοιχεία της πρότασης ε, είναι πολλά υποσχόμενα και είμαστε βεβαίως προσβλέπουμε στο να υπάρξει μια βαθιά συζήτηση συνεργασία βεβαίως με την ε, εισηγήτρια και όλους τους κοιόδους εισηγητές. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάνουμπαλ. Thank you. Um, Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μου δίνει τη δυνατότητα να συζητήσω και εγώ με τους συναδέλφου. τα σημαντικά αυτά ζητήματα. Θέλω να ευχαριστήσω την Τέρεσα Κομοντίνη για το έργο της, για την έκθεσή της. Πρέπει να πω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Είμαστε ήδη στις απαχές της όλης συζήτησης ε, και χαίρομαι που υπάρχει διαφάνεια και ανοιχτό πνεύμα. γιατί γνωρίζουμε ότι οι απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα θα είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Η ποια είναι η δική μου προοπτική κάτι που πρέπει από την οδηγία αυτή να εξασφαλιστεί είναι οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς, δημιουργοί, οι ερμηνευτές και όλοι όσοι εργάζονται στο πλαίσιο αυτού του μεγάλου φάσματος θα πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι από τα βασικά στοιχεία της οδηγίας. Έξω και είναι σημαντικό να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε πράγματα που μας έχουν τεθεί πολλές φορές, όπως είναι αυτή η διαφορά στην αμοιβή, αυτό το, το value gap και θα πρέπει να γίνει μια αναλυτική αξιολόγηση του διαδικτύου. Γιατί το διαδίκτυο είναι θέμα εδώ. Μέσω του διαδικτύου γίνονται τα πράγματα δεν χρειάζεται να αναλογικά έγγραφα ε, τα έργα. Ε, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το διαδίκτυο, γιατί πολύ περιεχόμενο είναι επιγραμμικό. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Άλλωστε το διαδίκτυο είναι σχετικά νέο ακόμη και κάπως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εν γέννη. Επίσης, ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, πρέπει επίσης να τα αντιμετωπίσουμε. Για τα νέα δικαιώματα των εκδοτών υπάρχει μια ε, διάταξη για περισσότερη δημιουργικότητα, περισσότερες επενδύσεις, ε, την υποστήριξη των δημιουργικών έργων και για μια διαφοροποιημένη ε, δημοσιογραφία. Αν όμως αυτό το θέμα, τα δικαιώματα των εκδοτών και το γενικότερο θέμα της δίκης αμοιβή δεν το έχουμε ως προτεραιότητα, θα δούμε ότι αυτό θα είναι πολύ επιζήμιο στις δημιουργικές βιομηχανίες, δημιουργικούς κλάδους, διότι γιατί να ασχοληθεί κανείς με αυτό το επάγγελμα, να γράφει, να παράγει έργα δημιουργικά, εφόσον δεν θα αμοιβέται επαρκώς. Αυτό είναι και το όλο θεμέλιο, κατ' εμέ, της οδηγίας και θα πρέπει να στηρίζει και όλες μας τις προτάσεις και διατάξεις. Επίσης, άλλες, σε σχέση με άλλες διατάξεις, για τους συνδέσμους, τα links, το έχουμε συζητήσει. Είναι ένα επικουρικό ε, πραγματικό δικαίωμα, αλλά τους ξέρουμε γιατί συζητούμε εδώ. Εν γέννη και το όλο θέμα των πλατφορμών γιατί σίγουρα η Google και άλλες μεγάλες πλατφόρμες είναι πολύ επιτυχημένες, έχουν να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Θα πρέπει όμως συγκεκριμένα ε, να ρυθμίσουμε τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ε, πλατφόρμων, γιατί αυτό το χάσμα, οι διάφορες αμοιβέ και τα προβλήματα τα σχετικά οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας αυτών των πλατφορμών σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει το ζήτημα αυτό να μας απασχολήσει. Οι πλατφόρμες πρέπει να αμείβουν τους δημιουργούς και τους ε, συγγραφείς και όλους τους ερμηνευτές με τον ε, ορθό τέρο δυνατό τρόπο και το σύστημα πρέπει να λειτουργεί επίσης με το τον τρόπο και προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης. Δεν θέλουμε όμως μόνο δημιουργικότητα από κάθε της μορφή, θέλουμε και μεγαλύτερη ποιότητα. Η παραγωγή του περιεχομένου είναι κάτι πολύ ε, σημαντικό και μπορεί να ε, υποβοηθηθεί από το διαδίκτυο με πολλούς τρόπους και αυτό είναι θετικό. Όμως θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την ποιότητα. Υπάρχουν λοιπόν μείζωνα ζητήματα που θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα τώρα να, καθίστε, να μειώσουμε τη συζήτηση, αλλά έχει πάει ήδη 10 παρά 20 και καλό θα ήταν να προσέχουμε και λίγο τι ώρα είναι. Έχουμε τρει ακόμα ομιλητέ, μετά θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή και μετά η Τερέ Κομωτίνη προφανώ θα επανέλθει για να κλείσουμε τον κατάλογο. Η κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, πολύ σύντομα, διότι μας πιέζει και ο χρόνος. Θα ήθελα απλώς ε, λίγο να συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφος η Μέρη Χάνιμπολ, να επανέλθω στην ουσία. Κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει ε, καθόλου να ε, φοβηθούμε με όλο αυτό το έργο της ε, μεταρρύθμισης των δικαιωμάτων του δημιουργού, το οποίο επιβάλλεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και από την εκβάθρων μετατροπή του τρόπου με τον οποίο οι συμπολίτε μας έρχονται σε επαφή με πληροφορίες και πολιτισμό. Η ουσία είναι να μην αποδυναμώσουμε ένα σύστημα, ένα οικοσύστημα το οποίο υποστηρίζει, προωθεί και χρηματοδοτεί τη δημιουργία, ε, την πολιτιστική δημιουργία που αποτελεί και τη βάση επί της οποίας ε, θα πρέπει ε, να συνεχίσει να ευημερεί η δημιουργική βιομηχανία και η πολιτιστική βιομηχανία με αξίες στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την εργασία, τη σωστή αμοιβή για την εργασία ε, και η επιβράβευση της αξίας κάποιου. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είχαμε την ευκαιρία να το πούμε αυτό. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την ε, ε, η την Τερέσκο Κομοντίνη, η οποία έχει ήδη κάνει πολλή δουλειά και μας απέδειξε ότι μπορεί να ε, κάνει πάρα πολλή δουλειά. στο άρθρο 13 που αφορά το θέμα του προστατευόμενου περιεχομένου και τις σχετικές αιτιολογικές σκέψεις που αφορούν το θέμα αυτό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τις διατάξεις του άρθρου 13 δεν ε, υπάρχει καμία περίπτωση να τη διαγράψουμε και να αποδυναμώσουμε ε, την ουσία αυτού του άρθρου. Πρέπει πραγματικά να έχουμε ως γνώμονα την ε, προτεραιότητα που μας εξωθεί να δοθεί νέα ισορροπία στην αμοιβέ των δημιουργών, διότι όλα όσα αφορούν τα θέματα των δημιουργών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν ε, μεγάλες πλατφόρμες οι οποίες αναδύονται, οι οποίες ε, έχουν και πάλι αναταρρήξει όλο το οικοσύστημα και δεν θα ήθελα να αρχίσουν να εμφανίζονται πάρα πολύ αμφιλεγόμενες θέσεις και να ερίζουν συνεχώς οι απόψεις, αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και το πόσο ευάλωτε μπορεί να γίνουν κάποιες διατάξει, οι οποίες στόχο έχουν ε, να ενισχύσουν κάποια πράγματα στην ψηφιακή εποχή και μπορεί να τα αποδυναμώσουν στην προσπάθεια αυτή. Και φυσικά υπάρχει και ε, πολύ ε, λογικά αντίστοιχο αίτημα από τους δημιουργίες. Αυτά. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ανοιχτή συζήτηση που έχει ε, οργανώσει αλλά και τις ακροάσεις που έχει οργανώσει και νομίζω ότι πράγματι αξίζει να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο εδώ στην Επιτροπή για να επεξεργαστούμε αυτό το θέμα με την δέουσα προσοχή. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, θεωρώ ότι η πρόταση Κομισιόν είναι ολοκληρωμένη και βάσει του οικοσυστήματος που ε, περιέγραψε μόλις η συνάδελφος. Ε, νομίζω λοιπόν από αυτή την άποψη ότι η πρόταση της Κομισιόν ε, μπορεί να τύχει της υποστήριξής μας αν και φυσικά θα χρειαστεί να ξεκαθαριστούν ορισμένα ζητήματα, ποιε ακριβώ είναι οι επιδιώξει και ποιε όχι τη Κομισιόν. Πάντω, ε, συνολικά θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι θετική. Και θέλω να αναδείξω κάποια ζητήματα. Άρθρο 11. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν την άποψη ότι θα έπρεπε να διαγραφεί. Εγώ πιστεύω ότι οι εκδότες ε, θα πρέπει στο, στην ψηφιακή εποχή να ενισχυθούν ως προς την διαπραγματευτική τους θέση και γι' αυτό δεν συμφωνώ ότι, με εκείνους που ισχυρίζονται ότι η, ο πλουραλισμός ε, ισούται με την δυνατότητα του οποιοδήποτε να δημοσιεύει οτιδήποτε στο ίντερνετ. Χρειαζόμαστε εκδότες οι οποίοι θα εξασφαλίζουν μια δομή, μια ταξινόμηση, μια αξιολόγηση του περιεχομένου που θα εξασφαλίζουν κάτι τέτοιο και νομίζω ότι αυτό από μόνο του ε, έχει ε, μεγάλη αξία και πρέπει ε, να δούμε πώς στην ψηφιακή εποχή θα εξασφαλίσουμε αυτόν τον ρόλο πώς θα δώσουμε τα εχέγγυα εκείνα που θα δώσουν ε, στους εκδότες τη δυνατότητα να επιτελέσουν το πολύ σημαντικό έργο τους. Ως προς, την, ε, προς το δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε, ε, είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις. Πάντως θέλω να πω ότι ε, η πρόταση Κομισιόν θα έρθει 14 έως 16, όπου γίνεται αναφορά στις συμβάσεις με τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς του περιεχομένου, αλλά και τις αμοιβέ αυτών, είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει ε, επί μακρόν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ε, ε, αμοιβέ δίκαιες για τους δημιουργούς. Και ένα γενικό θέμα θα ήθελα να θέσω. Τον Δεκέμβριο στην Ολομέλεια υπερψηφίσαμε μια έκθεση για, για το δημιουργικό περιεχόμενο και με αυτόν τον τρόπο ε, ε, τονίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει ε, πλούτο στον κλάδο των, της δημιουργικότητας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια ορθή κατανομή της αξίας του πλούτου που παράγεται μέσω του, των δημιουργικών ε, κλάδων, στο διαδίκτυο. Και από αυτή την άποψη λοιπόν η Κομισιόν ε, θεωρώ ότι έθεσε, υπέβαλε μια θετική πρόταση. Έχω και ένα ε, ερώτημα όσον αφορά τα snippets, τα links, τα hyperlinks. Εκεί αναφέρεται διαρκώς ότι θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ως προς το κείμενο που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει στο διαδίκτυο. Ε, χθες δημιουργήσαμε, ε, διοργανώσαμε ως πολιτική ομάδα και μια σχετική ακρόαση και εκεί διαπίστωσα με βάση και τις τοποθετήσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές σε αυτόν τον τομέα. Ακόμη και μετά την ε, έγκριση της πρώτης Κομισιόν θα μπορεί κανείς να δημιουργεί ε, υπερσυνδέσμους και θα ήθελα ε, αν μπορούσε η Κομισιόν να ξανατοποθετηθεί και να μας ε, εκθέσει για άλλη μια φορά ολοκληρωμένα τη θέση της. Ο κ. Καβαντά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την οδηγία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Διαπιστώνουμε ότι είναι ενδιαφέρον το κείμενο της Κομισιόν αλλά και η συνάδελφός μας η Τερέζα Κομωτίνη μας έχει ε, παρουσιάσει επίσης ε, μια πάρα πολύ καλή έκθεση διότι επικαιροποιεί τα ζητήματα που άπτονται των πνευματικών δικαιωμάτων σε συνάρτηση με την πρόοδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Θα ήθελα να κάνω στο δυνατόν και εγώ πιο γρήγορα κάποιε παρατηρήσει. Καταρχά, ποια είναι τα βασικά σημεία αυτή τη πρόταση οδηγία. Καταρχά, ε, υπάρχει ένα καλό νέο. Συγγενικά δικαιώματα για του εκδότε. Πολύ μεγάλη πρόοδο. Επίση, η υποχρέωση ε, αυτή σαφηνίζει κάπως την κατάσταση. Η πρόσβαση ελεύθερη ε, και η εύκολη δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχουν ε, έξοδα, δεν υπάρχει κόστος για κανέναν, άρα υπάρχει και η ανάγκη για υποχρέωση για δίκαιη αμοιβή και συμφωνώ και εγώ. Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, γιατί δεν θα πρέπει οι μικροί εκδότες ιδίως να τιμωρηθούν, οι οποίοι μάλιστα συμβάλλουν ενεργά στην ε, πολιτισμική ποικιλομορφία και πολλές ε, φορές ε, τα κείμενα τα οποία εκδίδουν είναι πάρα πολύ πρωτότυπα, αλλά τα μεγάλα σήματα δεν τα αναλαμβάνουν μεγάλες πλατφόρμες γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχουν, ότι θα έχουν απήχηση. Το άρθρο 13, το, το ξακοχάσμα βάλει gap, όλοι το ανέφεραν και σε αυτό θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Είναι σίγουρα κάτι από τα πλέον αναμενόμενα για τον πολιτισμικό κλάδο συνολικά. Οι πρακτικές ορισμένων επιγραμμικών πλατφορμών που παράγουν κέρδο, ε, διαδίδοντα περιεχόμενο προστατεύεται από το δίκτυο πνευματική ιδιοκτησία. αλλά χωρίς ταυτόχρονα ε, αυτήν την αξία να την κατανέμουν ε, ισομερός στους παραγωγούς είναι ανήθικο και μη φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτού του είδους την προσέγγιση αυτή, αυτόν τον τρόπο λειτουργίας γιατί κάθε προϊόν έχει την αξία του γιατί όχι αυτά λοιπόν. Η πρόταση της Κομισιόν είναι οι πλατφόρμες να έχουν ένα λογισμικό αναγνώρισης περιεχομένου. Με βάση το μοντέλο που ξέρουμε που χρησιμοποιεί το YouTube και που λειτουργεί. Και εκεί εντοπίζονται παραβιάσεις. Όμως, δεν φαίνεται απόλυτα θεμητό η δημιουργή οι εμπλεκόμενοι στο φορέα να έχουν ε, το δικαίωμα να παρεμβαίνουν ε, στο πώς εκμεταλλεύονται αυτά τα έργα οι πλατφόρμες. Δεν είναι θετική διάταξη, αλλά δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Οι δικαιούχοι σίγουρα έχουν ένα μοχλό διαπραγμάτευσης απέναντι στους γίγαντες του διαδικτύου, αλλά δεν ρυθμίζεται και εντελώς το ζήτημα της ευθύνη των επιγραμμικών πλατφορμών. Ε, για μένα ε, το θέμα είναι πολύ σημαντικό και θα το εξετάσω εκ του σύνεγγης. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εγγύψουμε στο ακαθόδε ζήτημα της ευθύνης των πλατφορμών. Δεν μπορούν ε, να προχωρούν έτσι σε χαρτογράφητα ύδατα. Επίσης ό,τι αφορά τα δικαιώματα δημιουργού για την επέκτασή τους ε, στην εξόριξη δεδομένων κειμένων data και text mining. Οι ερευνητές θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε αυτοματοποιημένες έρευνες πάνω σε αυτό το ακαδημαϊκό ε, ψηφιοποιημένο υλικό. Αυτό είναι δεδομένο και θα πρέπει με τη δική μας τη θέση να διευκολύνουμε τη δουλειά αυτών των ερευνητών. Συμφωνώ ότι οι διατάξεις επιτρέπουν στους ερευνητές να κάνουν έρευνες ε, μεγαλύτερη εμβέλειας πλέον. Όμως, για μια ακόμη φορά θεωρώ ότι αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να ε, τελειοποιηθούν για να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα ερευνητέ ε, ε, χωρίς ε, καμία, κανένα περιορισμό. Ναι, υπάρχει καινοτομία με την εξαίρεση αυτή, αλλά θα πρέπει η εξαίρεση να είναι πραγματικά εξαίρεση, άρα να οριοθετηθεί με το σωστό τρόπο. Ξέρουμε ότι ε, ο στόχος είναι ερευνητικοί οργανισμοί, αλλά αυτό είναι λίγο αόριστο στην ψηφιακή εποχή τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να διατηρηθούν και να μεταφερθούν στη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά χωρίς η πηγή δημιουργίας να καταστραφεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Καβαντά. Ζητώ τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δυνατόν σύντομα να παρέμβει. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα θα σας τα πω. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Καμα για τη δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε χθε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όπως υπόθηκε, βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια των συζητήσεών μας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διατηρήσουμε έναν έντονο ρυθμό προκειμένου να επεξεργαστούμε ε, το θέμα αυτό εντός της κοινοβουλευτική θητεία. και φυσικά δεν είναι η μοναδική πρόταση αυτή που συζητείτε Ταυτόχρονα προσπαθούμε να κλείσουμε τις συζητήσεις για τη φορητότητα. Ε, γνωρίζει και η κυρία Κομμοντίνη ότι μας ενδιαφέρει να προχωρήσουν αυτά τα δύο θέματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ε, και υπάρχει και ένα έργο στον τομέα των ευθυνών των ε, ραδιοτηλεπτικών οργανισμών. Τώρα, ως προς τις λεπτομέρειες της πρότασης, θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια σημαντικά ε, στοιχεία. Αναφέρθηκαν κάποια από αυτά και στις παρεμβάσεις των ε, βουλευτών. Φυσικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία ε, και κάθε ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής μας είναι να γίνονται σεβαστοί όλοι οι στόχοι πολιτικής στο πλαίσιο των πνευματικών ε, δικαιωμάτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι τι είδους ε, συζήτηση θα γίνει. Και δεν είναι καινούριο αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν τα, το, υπάρχει για παράδειγμα το θέμα των ε, εμπορικών διανομέων που θέλουν να χρησιμοποιούν τα πάντα ε, πληρώνοντας είτε πάρα πολύ λίγα χρήματα είτε και τίποτα. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά τα ε, τα δικαιώματα των δημιουργών. Πάντως τα επιχειρήματα που ακούγονται δεν είναι και πολύ καινοτόμα. Ε, όταν κανείς λέει ότι το διαδίκτυο είναι ένα καταπληκτικό μέσο για την ε, για την προαγωγή του έργου των δημιουργών. το ίδιο επιχείρημα είχαν χρησιμοποιήσει τη δεκαετία του 50 και οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν το, το περιεχόμενο δημιουργών χωρίς να τους αμείβουν. Ε, αυτό λοιπόν ε, πρέπει να το έχουμε κατά νου. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Πράγματι πρέπει να γίνει σε βάθος συζήτηση. Αλλά αυτό που χρειάζεται να μην ξεχνούμε και είναι ε, θεμελιώδες όσον αφορά τη συζήτηση για την ενιαία αγορά είναι πώς θα προωθήσουμε τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για έναν τομέα όπου έχει ε, επιλεγεί ένας δρόμος ε, μη εναρμόνισης. Ας το σκεφτούμε όμως. Η πραγματικότητα στα κράτη-μέλη. Ε, οι βιβλιοθήκες, τα εκπαιδευτικά συστήματα, η έρευνα στα διάφορα κράτη-μέλη παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διαφορές. Μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την λειτουργία λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ε, θεσπίζοντας ε, ε, στον ένα στον άλλο βαθμό ενιαίους κανόνες. Αν κάποιος έχει δουλέψει ποτέ στην έρευνα στην Γερμανία και στη Γαλλία θα, καταλά... θα ξέρει πολύ καλά πόσο ε, δύσκολο και ανεδαφικό είναι στην πραγματικότητα να ε, επιδιώξει κανείς πλήρη εναρμόνιση. Κατά τη γνώμη της Κομισιόν, να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα, το άρθρο 13 είναι απόλυτα συμβατό με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, δεν έχουμε κάνει καμία αλλαγή, ε, ούτε έρχεται σε αντίθεση η πρότασή μας με το άρθρο 15. Αλλά ε, θα έχουμε το χρόνο και την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όσον αφορά το ερώτημα της κυρίας Νίμπλερ για, για τα links και τους, ε, και, και τους εκδότες ε, και τις πλατφόρμες. Αυτό που προτείνουμε είναι να υπάρξει μια, μια νέα κατηγορία συγγενικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια η πρότασή μας αναφέρεται και στα, δύο, ε, στα δύο είδη δικαιωμάτων που είναι το δικαίωμα παραγωγής και το δικαίωμα κοινοποίησης στο κοινό δεν υπάρχει ε, πρόθεση να υπάρξει ένας νέος ορισμός ε, για τα δικαιώματα αυτά που ε, προτείνουμε να θεσπιστούν. Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το, με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Θα ισχύει για τους εκδότες ό,τι ισχύει για παράδειγμα για τους συντάκτες ή τους συγγραφείς. Όσον αφορά τα links λοιπόν δεν ε, ε, υπάρχει λόγος να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην πρόταση ε, αλλά σε αποφάσεις του, του δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δημιουργία αυτού του νέου δικαιώματος εκδότη δεν επηρεάζει τα υφιστάμενα δικαιώματα που έχει κατοχυρώσει με αποφάση του και το δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και σίγουρα θα επανέλθουμε. Αλλά Τερέ, θα ήθελα να σου ζητήσω να είσαι πάρα πολύ σύντομη γιατί έχουμε καθυστερήσει μισή ώρα και έχουμε ένα κατάλογο ψηφοφοριών 82 σελίδων. Σε παρακαλώ λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη να ευχαριστήσω όλους για τις απόψεις του σήμερα το πρωί και προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Μέρι. Η Μέρι Χάνιμπολ. Συγγνώμη, έχω ξεχάσει την κάρτα μου. Ζητώ συγγνώμη. Ε, Μπορούμε να ξεκινήσουμε. To take out my card. I hope that I have it with me. Colleagues, can we first make a test to... Συνάδελφοι, να κάνουμε μια δοκιμή, να δούμε πόσοι ψηφίζουν. So I open the test. Άρχεται. How many do we have? We have 20. 21 with Mary. And it's just this, um, plus 20. 21. Did everyone Uh, έχουμε 22, 23. Τώρα υπάρχει ένας περιττός. Τώρα έχουμε 20 μόνο. 20 άτομα ψηφίζουν. Okay, then we start uh, with the first. Uh, Μπορούμε να ξεκινήσουμε. the first report on uh, civil law. Η πρώτη έκθεση είναι για τους ε, κανόνες για τη ρομποτική. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 146 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, συγγνώμη, ΙΜΚΟ 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρα 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 159. Υπέρ. Συγγνώμη, ξεκίνησα από το κατά. Υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2.11 υπέρ. Against.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 6 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Να κάνουμε έναν έλεγχο αν θέλετε. Τραν 6. Επαλήθευση. Εσείς είστε κατά, οπότε καταγράφετε μια ψήφο κατά ακόμα. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. MV9, και εδώ έχω και μία προφορική τροπολογία, να προσθεθεί στον αριθμό των ατόμων που ε, βρίσκουν χρησιμότητα στη χρήση των ρομπών και τα άτομα με την αναπηρία. MV9 υπέρ, με την τροπολογία κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχή εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 11 υπέρ Επαλήθευση. Ήμκο 11. Εγκρίνεται. MV24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται εγκρίνεται, συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 275 υπέρ. Κατά. Πρέπει να γίνει επαλήθευση. Κυρία Χάνιμπολ είναι κατά, αλλά στο μεταξύ βρήκε και την κάρτα της προφορίας της. Απορρίπτεται λοιπόν. Η 276 αποσύρεται. 277. Τροπολογία 277 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 278 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 33 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συγγνώμη, πρώτο τμήμα εγκρίνεται, αλλά δεν είδαμε πηγαίνει κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές Πρέπει να γίνει παλήθευση. Δεύτερο τμήμα τη συμβαστικής τροπολογία 33. Εγκρίνεται. 295. υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. MV31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 302 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 27, εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Νόμιζα ότι περιλαμβανόταν στο συμβασμό, αλλά αυτή η παράγραφος ε, κάπου ξεχάστηκε. Αν συμφωνείτε λοιπόν με την προφορική τροπολογία, τότε μπορούμε να κάνουμε μία ψηφοφορία. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 323 υπέρ. 323.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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 346-347 ταυτίζονται υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 348 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 354 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 355 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 355. Projected. Απορρίπτεται. 356 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 357 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 358 υπέρ, κατά, αποχές επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 358. Rejected. Απορρίπτεται. 361 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 359 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 359. Εγκρίνεται. 362 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 364 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 366 καταπίπτει, άρα φτάνουμε στην προφορική τροπολογία 1. Πρόκειται για κείμενο του παρατήματος, το οποίο θέλουμε να ευθαγρονίσουμε με την ψηφοφορία για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Να ε, ορίζεται από Ευρωπαϊκό Οργανισμό σε περίπτωση που δημιουργηθεί τέτοιο οργανισμό, γιατί εμεί δεν ζητήσαμε απαραίτητο να υπάρξει ε, ίδρυση ενό τέτοιου οργανισμού. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη προφορική τροπολογία και αυτή έχει ε, ως στόχο να υπάρξει εφηγράμμιση με την παράγραφο για την ευθύνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 371 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για την τροπολογία 371 ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 372 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 373 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 375 και 376 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ας το υπαλληθεύσουμε ψηφίστε παρακαλώ για τις τροπολογίες 375 και 376 Adopted. Εγκρίνεται. 377 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 378 υπέρ, κατά, αποχές, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα για να είμαστε σίγουροι. Adopted. Εγκρίνεται. 379 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 380 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 381 υπέρ, κατά, αποχές, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Rejected. Απορρίπτεται. 382 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 383 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 385 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 386 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές 3 υπέρ κατά αποχές ας το δούμε ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Rejected. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 όχι. Τροπολογία 5 και 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία ήτρε B υπέρ ήτρε B υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Rejected. Απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά να ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε για την τροπολογία 16. Απορρίπτεται. NVB υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμκο D, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμκο E, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβεβαστική 51, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ενβι α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για την ετολογική σκέψη D εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία γιατί ε, καλύτερα να λέει ο εισηγητής να χρησιμοποιηθεί η φράση to be trained αντί για το think, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε ε, παρακαλώ για την τροπολογία 23. Ναι εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση. Για την 25 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Η σκέψη E και συγκεκριμένα τροπολογία 25. It is in grey and it is written false if um, a compromise 52 is adopted. Uh, compromise 52 has not been adopted, so we have to vote. Λοιπόν, η συμβαστική 52 δεν εγκρίθηκε, γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε όλες τις γκρίζες τροπολογίες που βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, 25. Ψηφίσαμε, εγκρίνεται. 26. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ για την 29 30. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31. Υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω. Να το επαληθεύσουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 31 ηλεκτρονικά. Rejected. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. MP9. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 35. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίθηκε λοιπόν η τροπολογία 40, οπότε περνάμε στην τροπολογία 45, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την τροπολογία 50. 50. 5-0. Τροπολογία του κύριου Μπούντα. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Τελευταία πρόταση. Τέλος πάντων. Η 15 δεν έχει εγκριθεί. Η συμβιβαστική. Τέλος πάντων. Απορρίπτεται όπως και αν έχει. Τροπολογία 51. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 54 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε. 66. Λείπει μια ψήφος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπι 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά χμ, αποχές να ελέγξουμε την 75 Rejected. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 77. Περνάμε στην 81, έτσι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ. Wasn't adopted. 75 was not adopted. I'm sorry. Yeah, sorry. Έκανα ένα λάθος, λέει η Πρόεδρος, επειδή δεν έγινε δεκτή 75, πρέπει να ψηφίσουμε όλε τι επόμενες. Την 76 την ψηφίσαμε, τώρα ψηφίσουμε την 77, υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται την 81 την ψηφίσαμε και απορρίφθηκε την 82 ψηφίσουμε υπέρ κατά Αποχές δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Να επαληθεύσουμε την 82 καλύτερα. Rejected. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην NV2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NVK υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 92 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε την 94. Απορρίφθηκε. Η 93 έγινε δεκτή που σημαίνει ότι καταπίπτει 95 και 96. Πηγαίνουμε σε 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 113, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 124, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμπιβαστική 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν β υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την τραν B, β. Projected. Um, the draft as a whole electron... Απορρίφθηκε ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης. Adopted εγκρίνεται. Δεν θέλω να συγχαρώ εαυτήν, θα συγχαρώ όλους όσους βοήθησαν να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ψηφοφορία. Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για πιβατικά πλοία, Ζωή μπερζεγό. Μία ψηφοφορία έχουμε. Όχι. Τροπολογία 2. Υπέρ. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης Μπερζερών. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα το σχέδιο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Λείπει μια ψήφος. Εγκρίθηκε συγχαρητήρια Ζωέλ. Επόμενη. Επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση Μπούντα. εκκοστικές υπηρεσίε. Λάβοντας υπόψη τις αλλαγές της πραγματικότητας αγοράς. Τροπολογία είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Κάποιος δεν ψηφίζει. Λείπει ένας. Ο κύριος ε, Μωρή. Μάλιστα. Να βγάλετε την κάρτα του παρακαλώ. Απορρίπτεται. Το πλοίο 102 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να επαληθεύσουμε την 108 παρακαλώ. Απορρίπτεται. 109 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Να ελέγξω. Τι σημαίνει αυτό, απορρίπτεται. Λοιπόν, Συμβιβαστική 13 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κάναμε ένα λάθος. Ξεχάσαμε μία τροπολογία να ψηφίσουμε. Ψηφίσαμε τη συμβαστική 13, αλλά προηγουμένως έπρεπε να είχαμε ψηφίσει την 113. Άρα γυρίζουμε λίγο πίσω και θέτω σε ψηφοφορία την 113 υπέρ. 113 πριν την συμβιβαστική 13. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Άρα πάμε τώρα στην τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 122 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 129 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολή 135 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 136 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 139 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ δεν βλέπω κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ την 140. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 145 υπέρ. Κατά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 Ελέγχουμε παρακαλώ. 151. Απορρίπτεται. Την 151 ψηφίσαμε. 151. Να επαναλάβουμε, μάλιστα. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 156 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε όμως να επαληθεύσουμε 158 απορρίφθηκε 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 πρόεδρος. Εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές 66. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 168 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 169 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 172 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 173 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 16C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 179 εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 και 183 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 184 υπέρ όχι καταπίπτει 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 16 D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 189 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 ε ή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ, κατά Αποχές ελέγχουμε παρακαλώ. Εγκρίνεται 196 περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 202 είναι πανομοιότητα. Η του τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά. Εγώ θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Απορρίπτεται. Συμβαστική το 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 211 ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 215 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 217 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 24 Rejected. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται.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 Πάμε στην 62. 62. Υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Rejected. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 και 68-69 όλες μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 80 υπέρ, Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω, μια επαλήθευση. Για την 80. Rejected. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. 81. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 δεν ψηφίσουμε. 8α συμβαστική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ναι, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σχέδιο γνωμοδότησης συνολικά ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπούντα. So, and now we come to the last... Και τώρα περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία. Το σχέδιο γνωμοδότησης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 44 επαλήθευση. Ε, Εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά. Πρέπει να το παληθεύσουμε γιατί δεν βλέπω κανέναν. 45 υπέρ. Συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Εφόσον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 Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη 55. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 59 59 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 59 εκρίνεται 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, όχι, 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά για την 66 Είμαστε στην 66. Τον κύριο Μπούντα κοιτάει, γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είμαστε στην 66. Ξαναπάμε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 και 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την 69. 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 72 και 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 73 και 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 86 δεν την ψηφίζουμε. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 80 η κυρία Ρέντα. Εκ μέρου του σκιώδης ηγητή μα του κ. Ντουράν, δεν δεχόμαστε την προφορική τροπολογία στην 89. Άρα ψηφίσουμε την 89 χωρί την προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ Τη τροπολογία 89 χωρί την προφορική τροπολογία. Χωρί προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 90 όχι, 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται.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 Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα η τελευταία ψηφοφορία. η δημοσιοποίηση των πληροφοριών από κάποιες επιχειρήσεις και θηγατρικές υπηρεσίες. Υπάρχει μία ψήφος μόνο. Α, συγγνώμη. Πρέπει να φύγω, ο κύριος Καβαντά θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου. Ζητώ συγγνώμη, διότι πρέπει να αποχωρήσω και να πάω σε άλλη συνεδρίαση που έχω να σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Καβαντά θα αναλάβει την Προεδρία και πρέπει να σας πω ότι εγώ εξαντλήθηκα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 25. Θα ζητήσουμε λοιπόν αμέσως τώρα την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω συντομία την νομική γνωμοδότηση Βέβαια, εφόσον εσείς ε, και τα μέλη της Επιτροπής σας έχετε οποιοδήποτε ερώτημα, είμαι στη διάθεσή σας. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αναφέρω ότι σύμφωνα με την ε, νομολογία του δικαστηρίου, η επιλογή της νομικής βάσης ε, δεν είναι θέμα δεκτικής ευχέρειας. Δεύτερον, η επιλογή της νομικής βάσης για μια νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες που θα μπορούσαν επίσης και δικαστικά να ε, αναθεωρηθούν, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο του μέτρου. Αυτή είναι η κλασική προσέγγιση του δικαστηρίου. Με βάση τώρα, μάλλον ε, σε σχέση με την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2013-34, κάθος 34, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την ετολική σκέψη 12 της εν λόγω πρότασης, που ξεκάθαρα αναφέρει ποιος είναι ο στόχος της προτινόμενης οδηγίας περισσότερη διαφάνεια και δημόσιος έλεγχος ε, του φόρου στο της εταιριών με προσαρμογή του νομικού πλαισίου. Το άρθρο 50, δάφιο 1 της Συνέχισης Εκλογής της Ευρωπαϊκής ε, δίνει τη νομική βάση. Με την, κανονική, την τακτική νομοθετική διαδικασία μπορούν να εγκρίνονται οδηγίες ε, για την ελευθερία κατάσταση σε σχέση με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τώρα, το εδάφιο 2 του ίδιου άρθρου περιλαμβάνει έναν όχι πλήρη κατάλογο των περιπτώσεων ε, για τις οποίες ισχύει αυτή η νομική βάση. Και για τους σκοπούς ε, της παρούσας το άρθρο 50. Εδάφιο 2 και σημείο G είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Αρκετέ οδηγίε εταιρικού δικαίου έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφο 1 με στόχο να προστατευτούν τα συμφέροντα των μελών και άλλων ακόμη και όταν αυτό ενέχει επαιτήσει αποκάλυψης πληροφοριών και ιδίω στη κοινή γνώμη. Παρομοίω, ο στόχο και το περιεχόμενο τη προηγούμενης οδηγία είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος δημόσιος έλεγχος των εταιρικών εσόδων και φόρων των πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εταιρείε αυτές, όταν έχουν συγκεκριμένο τζίρο, θα πρέπει, υποχρεούνται να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ετήσιες φορολογικές δηλώσεις. Άρα υπάρχει σύμφωνα με την πρόταση σχέση μεταξύ διαφάνεια και δημόσιου ελέγχου αφενός και συμφερόντων μελών και άλλων αφετέρου που είναι και ε, δικαιούχοι ε, και αυτοί που αποφελούνται των εγγύσεων που θα πρέπει να εγκριθούν δυνάμει του άρθρου 52G. Τώρα, οι όροι, μέλη και άλλοι. Αυτό αφορά το κοινό ευρεία Άρα όχι μόνο αυτούς που έχουν συμβατικές ή προσυμβατικές σχέσεις με μια εταιρεία και επηρεάζονται άμεσα από τις ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεύτερον, οι πρώτες πραγματικά υπηρετά συμφέροντα των ελόγων μελών και άλλων. Σύμφωνα λοιπόν με την ομολογία, αυτή είναι έννοια των άλλων λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο σε άτομα τα οποία έχουν άμεση συμβατική ή προσυμβατική σχέση με μια εταιρεία, όπως είναι οι πιστωτές για παράδειγμα. Όμως, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και ανταγωνιστές των εταιριών αυτό. Όπως επίσης το κοινό ευρύτερα. Η πρόταση λοιπόν βασίζεται στην υπόθεση ότι η δημοσιοποίηση πληροφοριών ε, για τον εταιρικό φόρο εισοδήματος συγκεκριμένων μεγάλων εταιριών προστατεύει τα συμφέροντα τα δημόσια συμφέροντα, τα συμφέροντα του κοινού που είναι και ο δικαιούχο ε, της συμμόρφωσης, μάλλον που είναι αυτός που αποφελείται από τη συμμόρφωση των εταιριών με τις διατάξεις ε, του φορολογική νομοθεσίας. Και με αυτό στόχο είναι να αποφευθεί και η μετατόπιση κερδών. Η διάθεση αυτών των πληροφοριών σε κάθε κράτο μέλος θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει έλεγχο της συμμόρφωση με τι φορολογικέ διατάξει και να γίνει επίσης και μια πολιτική συζήτηση για τα επίπεδα, τους συντελεστές αυτούς φορολογικούς και σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ένωσης. Επομένως αυτή η προστασία εμπίπτει και στο πλαίσιο του όρου συμφέροντα, interests, κατά την έννοια του 52G. Άρα συντονίζοντα το φυστάμενο νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει που επιβάλλονται στι εταιρείε και του κλάδου ε, σε σχέση και τα παραδείγματά του σε σχέση με την ε, δημοσιοποίηση φορολογικών πληροφοριών για την προστασία των συμφερόντων των μελών και άλλων, θεωρούμε ότι η πρόταση, ε, ο στόχο τη και το περιεχόμενο αντιστοιχούν στο άρθρο 50 τη συνθήκη για την λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει κάποια άλλη πιο συγκεκριμένη νομική βάση παρά μόνο το άρθρο 50 παράγραφο 1. Το όλο σύστημα γενικά της αναρμόνισης ε, της εσωτερικής αγοράς, άρθρα 114 και 115 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκειται ρητός σε άλλες νομικές βάσεις εφόσον αυτές υφίστανται. Αλλά αυτό δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως, το ότι υπάρχει το άρθρο 50,1 50, ε, ως η νομική βάση αποκλεί τα άρθρα 114 και 115. Και αυτή είναι οι λόγοι του οποίου η νομική υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το άρθρο 50, παράγραφο 1 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατάλληλη νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Euh. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ξεκάθαρες εξηγήσεις σας. Δεν ξέρω αν θέλει η Κομισιόν και το Συμβούλιο να παρέμει, το Συμβούλιο, ε, μάλλον η Κομισιόν πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν ε, επικροτεί τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία συμφωνούμε απολύτως. Δεν θα σας εκπλήσει άλλωστε εδώ στην Επιτροπή σας. Ε, η πρότασή μας ε, στόχο έχει να προωθήσουμε τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο. Ε, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την φορολογική νομοθεσία η πρότασή μα, είτε είναι ουσιαστική είτε διαδικαστική, δεν εναρμονίζει του φορολογικού κανόνε και δεν θέλει να εναρμονίσει το φορολογικό δίκαιο και να προστατεύσει τη φορολογική βάση των κρατών μελών. Και εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω επίση ότι έχουν εγκριθεί αντίστοιχε διατάξει ε, βάσει του άρθρου 50 ε, παράγραφος 1 στο παρελθόν για την εξορεκτική βιομηχανία και τη δασοκομεία και όλα αυτά έχουν γίνει βάσει του άρθρου 50 ε, παράγραφος 1 και δεν έχουν αμφισβητηθεί σε καμία περίπτωση. Επομένως, ε, τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε άλλη περίπτωση ότι οποιαδήποτε διάταξη η οποία τρόπον την να αναφέρεται σε θέματα διαφάνειας ε, φορολογικών απαιτήσεων θα πρέπει να βασίζονται στο άρθρο 115. Δεν μας φαίνεται ότι υποστηρίζεται και ότι υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Ε, άρα συμφωνούμε απολύτως και υποστηρίζουμε ε, τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο θέλει το λόγο. Η Προεδρία σημειώνει την νομική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και θα ε, αναφέρει το ζήτημα στα κράτη-μέλη. Η νομική γνωμοδότηση της ε, νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου δεν είναι η ίδια κατά την άποψή μας και η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εξεταστούν από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας... Α, συγγνώμη, η κυρία Ρέγνερ, δεν σας έβλεπα γιατί είστε ακριβώς εκεί που πέφτει το φως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο ερώτημα θέλω να απευθύνω στην Προεδρία. Ε, ποιος θα είναι ο ρυθμός, ποια θα είναι η ταχύτητα των εργασιών, πώς ε, δηλαδή θα εξελιχθεί το χρονοδιάγραμμα ε, το επόμενο διάστημα. The council, um, and the... Το Συμβούλιο και η Προεδρία θα χειριστούν τη διαδικασία αυτή με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Θα περιμένουμε τις εκθέσεις των Επιτροπών ΕΚΟΝ και Γιούρι και στο μεσοδιάστημα θα συνεδριάζουν και δικές μας ομάδες εργασίας προκειμένου να καταλήξουμε σε θέση των κρατών μελών και από εκεί και πέρα να ε, προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, καθώς και εσείς από πλευράς Κοινοβουλίου θα ολοκληρώνετε τη σύνταξη των δικών σας ε, εκθέσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση που είναι πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνη. και που κάθε άλλο παρά θετική είναι για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εδώ έχουμε μια διαφωνία ως προς τη νομική βάση ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό αντικατοπτρίζει και την συμμετοχή ε, των ε, συνομοθετών ε, κατά την νομοθετική διαδικασία. Το Κοινοβούλιο κανονικά θα έπρεπε να ε, προσφύγει στο δικαστήριο. Έτσι όπως έχουν δημορφωθεί τα πράγματα. Αυτές οι διαμάχες ως προς την, ε, τις αρμοδιότητες οδηγούν σε τραγέλαφο πολλές φορές. Και έχουμε να κάνουμε μια τέτοια περίπτωση. Και εδώ. Η διάσκεψη των Προέδρων επέλεξε δύο επιτροπές, δηλαδή την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, και εμείς θεωρούσαμε ότι ενέπιπτε το θέμα αυτό στην αποκλειστική μας αρμοδιότητα και την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Έχω διάφορες παρατηρήσεις να κάνω για το CCC και του τους ε, υπαλλήλους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το συζητήσουμε σήμερα αυτό, θα το συζητήσουμε στις συνεδρίες των συντονιστών. Θέλω πάντως να αναφέρω ότι οι φορολογικέ υποθέσεις ε, ε, αποτελούν μεγάλο τμήμα των, ε, της, της εν λόγω πρότασης και γι' αυτόν τον λόγο ε, χρειαζόμαστε και την γνωμοδότηση, εν πάση περιπτώσει την εμπλοκή και της ε, ΕΚΟΝ. Ε, εγώ διαφωνώ και θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή όλων ώστε να μην επαναληφθεί άλλο τέτοιο λάθος. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Να σας πω ότι την άποψή μου. Να σας πω ότι εγώ συμφωνώ με την άποψη που εξέφρασε η νομική υπηρεσία και επιβεβαίωσε τα άλλα θεσμικά όργανα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τη σωστή επιλογή απόλυτα ορθή. Και όπως επεσήμανε και η νομική υπηρεσία, ο στόχος ε, της πρότασης, αφέστατα, είναι η αύξηση της διαφάνειας και ε, του δημοσίου ελέγχου των ε, φορολογικών εσόδων κάποιων επιχειρήσεων. Το στόχο, λοιπόν, έχουμε να τις ενθαρρύνουμε να υποχρεώνονται να ε, διαβιβάζουν τις απαραίτητες ε, πληροφορίες για τον ε, φόρο στις χώρες στις οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους. Ο φορολογικός στόχος λοιπόν της πρότασης είναι δευτερεύον και δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε αλλαγή της νομικής βάσης και κατά συνέπεια της νομοθετικής διαδικασίας η οποία θα προκύψει. Γι' αυτό και ακριβώς το άρθρο 50 της, Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κατάλληλο άρθρο. Ευχαριστώ. Προτείνω να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα για το θέμα αυτό. Ποιο είναι υπέρ τη πρόταση αυτή. Α, πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, συγγνώμη. Να μην υπάρχει καμία σύγχυση λοιπόν επί του ζητήματος. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσατε να μας πείτε συγκεκριμένα τι ψηφίζουμε, γιατί εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να ψηφίσω. Τη νομική βάση. Δηλαδή, να παραμείνει ε, το άρθρο 50 ως νομική βάση. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Est-ce que tout le monde a voté Ah. Allez-y, allez-y tranquillement. Ναι, με την ησυχία σα. Εξακολουθεί να λείπει ένα. Κάποιο δεν ψήφισε. Όχι, κάποιο λείπει. Πέρασε ψηφοφορία. Κανείς δεν είναι κατά, μία αποχή και δέκα υπέρ. Επομένως εγκρίνεται. Σχεδόν ομόφωνα και σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η συζήτηση αυτή θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, επομένως όσοι δεν ε, είναι ε, εξουσιοδοτημένοι να παραμείνουν, θα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Διακόπτουμε για ένα λεπτό για να αποχωρήσουν όσοι δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εδώ και θα συνεχίσουμε.